Καλημέρα, καθίστε για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Allora, noi continuiamo oggi la... Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα με την ε, συνεδρίασή μας ε, στις συζητήσεις του πρώτου κλάστερ για την διατήρηση των προσωπικών δεδομένων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, στην καταπολέμηση του οργανωμένου ε, εγκλήματος ε, και του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Εγκλήματος και τις διαδικαστικές εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ακούσουμε λοιπόν τη Σόφη Γκουάνσνη που είναι επικεφαλής του Τμήματος Προστασίας Δεδομένων του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα μας μιλήσει για την προάσπιση των δικαιωμάτων και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στο Σκοτ Κρόσμπι, ο οποίος είναι δικηγόρος ε, του Ευρωπαϊκού ε, Συλλόγου Δικηγόρων, που θα μιλήσει για τα ατομικά δικαιώματα στις ε, διασυνοριακές υποθέσεις. 15 λεπτά ο χρόνος ομιλίας για τον κάθε ομιλητή και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η συζήτηση και θα δοθεί χρόνος 2 λεπτά σε κάθε συνάδελφο να δώσω λοιπόν ε, καταρχάς ε, το λόγο στην ε, Σόφη Κουάσνη, επικεφαλής του Τμήματος Προστασίας Δεδομένων και να σας πω το εξής, εγώ θα φύγω στις 11 παρατέταρτο, θα αναλάβει ο κύριος Ρούι Ταβάρες ή ο κύριος Νιούτον Ντάνς Ταϊνία και η ακρόαση με την κυρία Βασιλιάδου αναβλήθηκε και η γραμματεία θα σας ενημερώσει πότε θα γίνει η νέα ακρόαση. Από τι 11 παρατέταρτο και μετά λοιπόν θα προεδρεύει είτε ο κύριο Ταβάρε είτε ο κύριο Νιούτον Ντάν. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σόφη Κουάσνη για ένα τέταρτο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλημέρα κυρίες και κύριοι σας, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είναι για μένα μεγάλη χαρά για το Συμβούλιο της Ευρώπης δηλαδή που συμβάλλουμε έτσι στις εργασίες σας και θα σας παρουσιάσουμε και τις δικές μας. Το σημερινό μας θέμα, η παρουσίασή μου δηλαδή, αφορά το δικαίωμα σε ιδιωτική ζωή και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αρχίζω δηλώνοντα ότι είναι σημαντικό για τις κοινωνίες μας να προστατεύονται και να καταπολεμάται το έγκλημα αλλά και να προστατεύονται οι θεμελιώδεις και ατομικές ελευθερίες ιδιαίτερα εκείνες που προβλέπονται από τη χάρτα των θεμελιωδών. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πλήρης σεβασμός και του νόμου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στην πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος υπάρχει τίθεται ένα θέμα προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων όπως περιουσίας, περίθαλψης και ιδιωτικής ζωής. Γενικά η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προστατεύει άτομα κατά αυθαιρεσιών και κατά μέτρων που το κράτος λαμβάνει γιατί πρέπει πάντοτε να αποκλείεται η αυθαιρεσία και η άνηση η ρατσιστική μεταχείριση. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που θα λαμβάνουν τα κράτη είναι νόμιμα, τα προβλέπει ο νόμος και όταν υπάρχει περιορισμός μερικών των δικαιωμάτων που χορηγεί η σύμβαση, τότε οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να ορίζονται ως εξαιρέσεις και προσωρινές εξαιρέσεις. Πρέπει δε να είναι αναλογικές με τον στόχο που στοχεύεται και απαγορεύεται η... απαγορεύονται τα βασανιστήρια, η προφυλάκηση έχει συγκεκριμένα όρια κτλ. Ιδιαίτερα το δικαίωμα για, στην ιδιωτική ζωή που είναι το άρθρο 8 της Συνθήκης των Δικαιωμάτων προβλέπεται με δύο παραγράφους. Η πρώτη μιλάει για το δικαίωμα του καθενός να έχει ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και η δεύτερη παράγραφος μιλάει για την πιθανή παρεμβολή των αρχών και περιορισμό του δικαιώματο αυτού εφόσον μόνο είναι απαραίτητο αυτό για τη δημοκρατική ζωή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και όπως σας είπα πρόκειται για εξαίρεση και γι' αυτό περιορίζεται και χρονικά. Η σύμβαση αναφέρει τις συνθήκες όπου επιτρέπεται αυτό. Εθνική ασφάλεια, δημόσια ασφάλεια, οικονομική ευημερία του κράτους, ε, προστασία της τάξης ή ε, προστασία της ελευθερίας άλλων. Οι περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό παίρνουν διάφορες μορφές. Μπορεί να αφορά θέματα όπως σωματική έρευνα, οικιακή έρευνα, μυστικές υπηρεσίες κλπ. Δεν ορίζει η σύμβαση βέβαια τι είναι η ιδιωτική ζωή, γιατί η έννοια αυτή έχει εξελιχθεί από την ομολογία του δικαστηρίου ιδιαίτερα. Ένα μεγάλο τμήμα της είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το δικαστήριο πολλές φορές έχει πει ότι και μόνο το γεγονός της καταχώρησης προσωπικών πληροφοριών είναι παρεμβολή και περιορισμός του δικαιώματος σε ιδιωτική ζωή. Επομένως τίθεται το ερώτημα ικανοποιούμε τις συνθήκες του παραγράφου 2 του άρθρου 8. Η ίδια η συνθήκη δεν αναφέρεται ρητά στο δικαίωμα στην προστασία δεδομένων. Γι' αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης στις αρχές της δεκαετίας του 80 πρόσθεσε κάτι στη Σύμβαση για την προστασία των ατόμων ως προς τη χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων. Εγώ θα μιλήσω όμως μόνο για τα άτομα, γιατί αν και μιλάμε για προστασία δεδομένων, βασικά εννοούμε προστασία των ατόμων. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δικαίωμα του ανθρώπου μάλλον δηλαδή του ατόμου. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει χωριστή τέτοια διάταξη είναι γιατί πριν από 60 χρόνια όταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε συγγραφεί η έννοια της προστασίας των δεδομένων δεν υπήρχε ακόμα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιορίζεται στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ για το θέμα της, προστα... το... θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι καθολικό. Πριν από 30 χρόνια η σύμβαση προβλεπόταν για οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όχι μόνο για τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η σύμβαση αυτή η λεγόμενη 108 εξυγχρονίζεται αυτή τη στιγμή και υπάρχει εδώ ένας παραλληλισμός με αυτά που κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση την αναθεώρηση δηλαδή του νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων. Και τα δύο αυτά γίνονται σε συνεννόηση. Ξέρουμε τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες και Θέλουμε να είναι συμβατές οι δύο μεταρρυθμίσεις. Η Σύμβαση 108 έχει εγκριθεί από τα κράτη-μέλη της Ένωσης πάντως. Η Σύμβαση 108 αφορά και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι οριζόντια δηλαδή, έχει οριζόντιο εύρος. Αυτή είναι μια από τις ιδιαιτερότητές της. Η δημόσιος τομέα σημαίνει βέβαια επιβολή νόμου και τάξεως οι αρχές της είναι γενικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, η συλλογή να γίνεται νομοτύπος και η διεκπαιρέωση, τα δεδομένα να καταχωρούνται για θεμιτούς και νόμιμους λόγους, όχι για λόγους που δεν προβλέπονται από αυτήν, ούτε να κατούνται για χρόνο περισσότερο από όσον προβλέπεται. Επίσης, η ποιότητά τους πρέπει να είναι τα δεδομένα επαρκή σχετικά, όχι υπερβολικά, σε σχέση με το στόχο δηλαδή της διεκπαιρέωσης, ακριβή και τα άτομα που αφορούν έχουν ορισμένα δικαιώματα ως προς την πρόσβαση τους και διόρθωση στα δεδομένα. Εκτός από αυτές τις εγγυήσει για τη συλλογή και διεκπαιρέωση χρήση των δεδομένων, η Σύμβαση επίσης μιλάει για τα λεγόμενα ευαίσθητα δεδομένα ιδιαίτερη κατηγορία τους δηλαδή που χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία μεταξύ τους αυτών των ειδικών δεδομένων είναι και τα ποινικά μητρώα οι περιορισμοί στα δικαιώματα που ανέφερα επίσης προβλέπονται στη Σύμβαση 108 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο άρθρο 8 της. Οι περιορισμοί αυτοί είναι δυνατόν να επιβληθούν αν είναι περιορισμένοι, τελείως απαραίτητοι και σε μικρό αριθμό περιπτώσεων, δηλαδή δημόσια ασφάλεια, εθνική ασφάλεια και καταπολέμηση εγκλήματος. Παρακολουθούμε λοιπόν, βλέπετε, την ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως προς τους πιθανούς δυνατούς περιορισμούς. Αυτή λοιπόν είναι η λογική που ακολουθεί το δικαστήριο. Το δικαστήριο καθορίζει τρεις όρους με βάση τους οποίους μπορεί να επιβληθούν περιορισμοί στο δικαίωμα ιδιωτικής ζωής. Να είναι νόμιμο, να έχει θεμητό και νόμιμο στόχο και να εφαρμόζεται με δημοκρατικό τρόπο. Ο περιορισμός του δικαιώματος στην, ελεύθερη στην ιδιωτική ζωή πρέπει να είναι αναλογικός με το στόχο και οι λόγοι που εκθήθενται από τις δημόσιες αρχές για να δικαιολογήσουν το μέτρο αυτό πρέπει να είναι επαρκής. Οι όροι λοιπόν δεν μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα για όλες τις χώρες, αλλά το δικαστήριο κάθε φορά θα τις καθορίζει ανάλογα με την περίπτωση σε κάθε χώρα. κάθε χώρα. Τώρα, επίσης πρέπει να τονίσω ότι αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να συμφωνούν με τον νόμο. for by law. Δηλαδή να προβλέπονται και από τον νόμο. Ακριβώς για να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες. Πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα για τον ενδιαφερόμενο. Να έχει δικαίωμα δηλαδή να δει τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται και να είναι η όρη της πρόσβασης εύληπτη και ρητή. Η Σύμβαση 108 έχει γενικό εύρος όπως σας είπα, καλύπτει και το δημόσιο τομέα δηλαδή την επιβολή νόμου και τάξεως, αλλά είναι διατυπωμένη με πολύ γενικό τρόπο για να μπορεί να εγκριθεί από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης στα τέλη της δεκαετίας του 80 συνειδητοποίησε ότι μερικά μέλη του θεωρούσαν ότι το άρθρο 9 για τις εξαιρέσεις επέτρεπε στις αστυνομικές αρχές να μην εφαρμόζουν τις αρχές. Και το 87 η Επιτροπή Υπουργών νομοθέτησε περισσότερο τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από την αστυνομία σε εκείνο το κείμενο ισχύει ακόμη, δεν έχει απαρχαιωθεί και έχει συμπεριληφθεί στο κοινοτικό κεκτημένο μέσω της σύμβασης του Σένιγκεν. Και η τωρινή οδηγία που εξετάζεται για την ε, προστασία των δεδομένων έχει βασιστεί εν μέρη και σε αυτό. Τώρα θα ήθελα να κάνω μία σύνδεση με τη, μεταξύ της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Έχουμε και γι' αυτό μια σύμβαση που λέγεται Σύμβαση της Βουδαπέστης η οποία έχει ένα άρθρο 15 για τους όρους για τις εγγυήσεις που προβλέπει. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το κείμενο θα προστατεύουν επαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες καθώς μεταξύ των οποίων και όλα όσα έχει συνυπογράψει και προβλέψει η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Ευρώπης γνωρίζει πολύ καλά ότι οι συνυπογράφοντες πρέπει να προβλέπουν στην εθνική τους νομοθεσία και ένα κεφάλαιο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Άλλο σημαντικό άρθρο της σύμβασης αυτής για το κυβερνοέγκλημα αφορά την καταχώρηση των δεδομένων, τη διατήρησή τους. Αυτό το σκέφτονται και στην Ένωση αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιείται ως ορολογία η κατακράτηση δεδομένων, καταχώρηση, αποθήκευση. Η διατήρηση των δεδομένων αφορά συγκεκριμένο πλαίσιο καταπολέμησης του εγκλήματος και όχι δεν πρόκειται για γενική διάταξη και ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων περιορίζεται σε 90 μέρες, πολύ μικρός χρόνος. Τέλος, τονίζω ότι για το Συμβούλιο της Ευρώπης τα δικαιώματα που χορηγούνται από τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη προστασία των δεδομένων, στη Σύμβαση 108 δηλαδή, όλα αυτά τα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά και online και offline που λέμε. Έτσι προσπαθούμε να εγγυηθούμε ότι επειδή γίνονται πολλά στο ίντερνετ και υπάρχουν και θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και, και στο ίντερνετ να προβλέπονται και αυτά. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρόσμπι. Παρακαλώ. Uh, Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ πέρα. Και ελπίζω στο λίγο χρόνο που έχουμε να μπορέσω να συνεισφέρω και εγώ κάτι στην επίτευξη των στόχων σας. Το θέμα το οποίο πρέπει να αναπτύξω είναι πως τα ατομικά δικαιώματα ε, διασφαλίζονται σε διασυνοριακές διώξεις. Αυτό το οποίο θα τονίσω βέβαια είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τις ε, απόψεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Συλλόγου, ούτε κάνουμε τις απόψεις των συνεταίρων μου στο δικηγορικό μου γραφείο. Τούτου λεχθέντος τι εννοούμε ατομικά δικαιώματα. Λοιπόν, να το. για την παρουσίασή μας σήμερα. Ορίζουμε τα ατομικά δικαιώματα στα δικαιώματα σε δίκαιη δίκη. Αναφέρθηκε ήδη πριν από λίγο πως το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη διασφαλίζεται από το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και τα Σα καταπλήξει ίσως, ίσως και όχι, αλλά τα στατιστικά στοιχεία του δικαστηρίου δείχνουν πως από το 1959 μέχρι το 2011 υπήρξαν 8.482 ε, καταδίκες κρατών μελών της συνθήκης για μη σεβασμό των ε, δικονομικών δικαιωμάτων ε, πολιτών. Και αυτό σημαίνει 3.672 ουσιαστικέ παραβιάσεις των δικαιωμάτων και 4.810 παραβιάσεις της, του εύλογου χρονικού διαστήματος. Και βέβαια όλα αυτά ξεκίνησαν και όλα αυτά είναι απλά η κορφή του παγόβουνου και πρέπει να ξέρουμε πως ε, όσο περνά τα χρόνια συνεχίζουν τα καρτιμέλη να παραβιάζουν τα δικαιώματα αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό γιατί όσο περισσότερο παραβιάζεται τόσο ε, λιγότερο θεωρείται το σύστημα των πυρικών δικαστηρίων ότι έχει νομοποίηση και βεβαίω αυτό σημαίνει πως ε, και οι εισαγγελίες θα έχουν ε, επαρκής εξή, αλλά θα προστατεύονται και τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Και βεβαίω θα μιλάμε για διακρατικέ τέτοιε υποθέσει. υπάρχουν περισσότερε πιθανότητε παραποίηση αυτών των δικαιωμάτων για διάφορους λόγους. Παραδείγματο χάρη οι διασυνοριακέ έρευνε καθυστερούν ε, την υπόθεση. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο να διερευνηθούν ε, τα εγκλήματα αν υπάρχει διασυνοριακό στοιχείο. Όσον αφορά τον κατηγορούμενο ή τον ύποπτο, αυτός ή αυτή μπορεί να έχει δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στους μάρτυρες. Ε, τίθενται στήματα μετά για το πώς ε, χρησιμοποιούνται δεδομένα που έχουν ε, συλλεγεί στο κράτος Α, πώς χρησιμοποιούνται στην δίκη στο κράτος Β. Πάρα πολλά έχουν γραφτεί και δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω είναι να παρουσιάσω κάποιες πιθανές δυσκολίες με το να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Η υπόθεση αυτή, ας την πούμε JD, ε, εναντίον του Βελγίου, αφορούσε ακριβώς ένα δικονομικό ζήτημα ο JD λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εργαζόταν για μια εγκληματική οργάνωση στη Μάλαγα, στην Ισπανία όπου από το ότι φαίνεται υπάρχουν πολλές τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις. Είχαμε λοιπόν εδώ πέρα αυτό το οποίο ονομάζουμε μια απάτη σε πολλές ε, επικράτειες. Τι σημαίνει αυτό. Είναι η απάτη ήταν η εξής. Ομάδες ανθρώπων τηλεφωνούσαν σε πιθανά θύματα και τους ε, προσέφεραν ε, ε, οικονομικές υπηρεσίες ή κέρδος. Αυτό το οποίο τους προσέφεραν εδώ πέρα ήταν πωλήσει μετοχών σε εταιρείε σε που δεν υπήρχαν. σε επενδυτέ σε κάθε κράτος μέλος της Ένωσης και γνωρίζουμε πως η ε, συγκεκριμένη αυτή απάτη κράτησε πάρα πολλά χρόνια και κατάφερε να αφαιρέσει γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ από διαφορούς επενδυτές τα... Είχαν ξεκινήσει από τις ΗΠΑ, εκεί πέρα πήγαν τα λεφτά, οι άνθρωποι από τις ΕΠΑ δεν εκδόθηκαν. Αυτοί οι οποίοι συνέχιζαν ήταν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στις ΗΠΑ, δηλαδή ο πελάτης μου. ο οποίος παραδόθηκε, εκδόθηκε δηλαδή στη Γερμανία με βάση ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δικάστηκε, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε. Μόλις ε, αποφυλακίστηκε πήγε στην Ισπανία. Μετά από δύο-τρεις εβδομάδες έφτασε ένα ένταλμα σύλληψης από το Βέλγιο. Τον συνέλαβαν, τον πάνε στη Μαδρίτη, βρίσκεται ενώπιον ενός δικαστή και τελικά τον εκδίδουν στο Βέλγιο παρά το ότι ε, είπε πως είχε ήδη καταδικαστεί για αυτή την υπόθεση και φυλακιστεί. Αυτό το αγνόησαν οι Ισπανικές αρχές, τον στείλανε στο Βέλγιο, στο Βέλγιο είπε το ίδιο πράγμα, ναι είναι in idem, ότι κανείς δεν μπορεί να δικάζεται δύο φορές για το ίδιο πράγμα, για να μην τον κατηγορήσουν στο Βέλγιο, το αγνόησαν αυτό, γιατί, γιατί είχε καταδικαστεί για τελεσμένη απάτη στη Γερμανία, ενώ στην, ε, στο Βέλγιο ήθελαν να το δικάσουν για συνωμοσία. Αρνήθηκαν να τον ε, αποφυλακίσουν γιατί δεν ήταν ε, Βέλγος πολίτης αλλά κάτοχος Βρετανικού διαβατηρίου είχε προφυλακιστεί για 12 μήνες και μετά ε, ήθελε και η Φιλανδία αφού ε, δίκαζόταν και καταδικαζόταν πιθανώ ε, και αποφυλακιζόταν από το Βέλγιο, να τον δικάσει και εκείνη. Και βεβαίω το θέμα ήταν που θα πήγαινε αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, οι δυσκολίε αυτέ ε, έπρεπε να αποφεύγονται μέσω του συντονισμού της ε, Eurojust. Η Eurojust βεβαίως δεν έχει αρμοδιότητα για να κρίνει το ζήτημα αυτό ακριβώς των πολλαπλών δικαιοδοσιών, αλλά θα πρέπει να προλαμβάνει τέτοιες καταστάσεις και να με συγχωρείτε, ξέχασα εδώ πέρα τα τις Και, όπως είχε πει και ο Αντρέ Κλίπ, που είναι αυθεντία στο θέμα του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου πως η Eurojust θα έπρεπε να προλαμβάνει τέτοιες συγκρούσεις μεταξύ δικαιοδοσιών, πολλαπλών δικαιοδοσιών και ζητήματα νίδων. Θα έπρεπε να χρησιμοποιείται συχνότερα. Για να επανέλθουμε στην υπόθεση λοιπόν του πελάτη μου, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία νομίζω ενδιαφέρουν της, ε, τη συζήτηση της Επιτροπής σας. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν, ο JD εφόσον είχε φυλακιστεί ήδη στην Γερμανία για απάτη, γιατί εκδόθηκε στο Βέλγιο για να δικαστεί για το ίδιο δίκημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως την περίπτωση Χίκη παραδείγματος χάρη, έγινε δεκτό το Nebis in Eden ε, στο Βέλγιο. Ο άνθρωπος είχε φυλακιστεί στην ε, Γαλλία. Μόλις ε, αποφυλακίστηκε τον συνέλαβε το Βέλγιο, επικαλέστηκε τον Nebis in Eden και τον αποφυλάκησαν σε 10, σε μέρες. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτής της υπόθεσης και της υπόθεσης του JD στην υπόθεση Χίκη. Δεν υπήρχε... Υπήρχε ενάγων Δηλαδή κάποιος ο οποίος ε, είπε πως ήταν ε, θύμα της απάτης και ήθελε να αποζημιωθεί. Αυτός προσεύχε λοιπόν στις βελγικές αρχές και με βάση αυτή η προσφυγή εκδόθηκε ένα ευρωπαϊκό εντέλμα σύλληψης και ε, άρα Και άρα εκδόθηκε στο Βελγίο. Γι' αυτό ε, αρνήθηκαν να, να δεχτούν το ότι δεν μπορούσε να δικαστεί δύο φορές για το ίδιο πράγμα. Αλλιώς βεβαίω θα είχε απορριφθεί το αίτημα του ε, ενάγοντος. Ένα άλλο ζήτημα. Εάν ε, μπορούσαν όντως να του αρνηθούν το Nebis in idem, θα έλεγα όχι, γιατί εφόσον είχε ήδη καταδικαστεί και φυλακιστεί για την απάτη, την τετελεσμένη, δεν μπορούσε να δικαστεί και να καταδικαστεί για την απόπειρα μετά απάτης, γιατί αν έχει καταδικαστεί για ένα έγκλημα που έχει τελεστεί ήδη, η καταδίκη για την ε, απόπειρα ή την προπαρασκευή είναι πάλι καταδίκη για το ίδιο πράγμα. Και αυτό απαγορεύεται. Από το διεθνές δίκαιο, από την ΕΣΔΑ κτλ. Το επόμενο ερώτημα είναι γιατί κράτησε τόσο προφυλάκηση Η απάντηση είναι ε, το πως ε, τα προβλήματα με το διαβατήριο ήταν πρόσχημα γιατί τελικά ε, τον έβγαλαν με εγγύηση απλά τον προφυλάκησαν μόνο και μόνο για να ικανοποιηθεί ο ενάγων. Οπότε παρά το ότι είχε καταδικαστεί, δεν αμφισβητεί κανεί την ενοχή του. Είχε καταδικαστεί, έτσι. Ήταν ένοχο και, και την ποινή του. Αλλά το σύστημα είναι τέτοιο, ώστε κινδύνευε να περάσει την υπόλοιπη ζωή του ε, από τη μία χώρα στην άλλη, δικαζόμενος. Σε όσες χώρες είχε ξαπατήσει ανθρώπους. Τι σχέση έχει αυτό με τη δουλειά της Επιτροπής σας. Προσπαθώ να σας πω πως σε μια Ευρώπη 27 καρτών μελών 28 δηλαδή με 28 συστήματα ποινικού δικαίου υπάρχουν πάρα πολλές ε, διαφορές ε, ασυνέπειες παραδείγματος χάρη η έννοια του ενάγοντος δεν υπάρχει σε πολλά νομικά συστήματα και θεωρείται, μάλιστα σε ορισμένα από αυτά, πως η παρουσία του ε, διαταράσει την διαδικασία της ε, ποινική δίκης. Αλλού στην Ένωση είναι ε, πλήρως αποδεκτό. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα μια σύγκριση. Το Nebis in Idem είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Ιδεωδός θα έπρεπε να αποτρέπει την έκδοση από το ένα κράτος ε, στο άλλο, όπως ε, αναφέρει το άρθρο 3 του Ευρωπαϊκού ε, Εντάλματος Σύλληψης. Αλλά στην πράξη δεν γίνεται αυτό. Ένα άλλο ζήτημα. Είναι πως ιδεοδός το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα έπρεπε να μπορεί να διορθώνει τέτοιες ε, καταστάσεις. Αλλά τι συμβαίνει, είναι τόσο υπερφορτωμένο το δικαστήριο, ώστε μόνο 5% των υποθέσεων που φτάνουν στο δικαστήριο, φτάνουν στο ακροατήριο τελικά. Οπότε, Τι έχουμε, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σύστημα ποινικού δικαίου που λειτουργεί με βάση την αμοιβαία αναγνώριση, αλλά τελικά μέσα σε αυτό το σύστημα υπάρχουν τόσο πολλά αντιφατικά στοιχεία, ώστε ο κίνδυνος ε, παραβίασης ε, του δικαιώματος ε, δίκαιη δίκη είναι πάρα πολύ υψηλός, ειδικά σε περιπτώσεις με τρίτα κράτη. Θα χρειαστεί όντω, θα χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνος για να ε, μην υπάρχουν ε, αντιφάσεις στο σύστημα εντό τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Η γρηγορότερη λύση θα ήταν να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να υπάρξει ένας ομοσπονδιακός Ευρωπαϊκός Ποινικός Κώδικας. Έτσι και η ε, η εισαγγελία θα μπορούσε να ωφεληθεί και βεβαίως ε, η υπεράσπιση γιατί θα ήταν βεβαίως ε, ευκολότερη και η πρόσβαση στα στοιχεία και στους ε, <laughs> μάρτυρες και το πρόβλημα το οποίο περιέγραψα με τις πολλαπλές ε, δικαιοδοσίες δεν θα υπήρχε. Νομίζω ο χρόνος μου τελειώνει. Ίσως τα δύο, αν μου δίνετε τα δύο λεπτά τα οποία δεν μίλησε, στα οποία δεν μίλησε η προηγούμενη μιλήτρια. Κοιτάξτε, το, αυτό το οποίο σας ανέφερα ε, δεν είναι πάρα πολύ δημοφιλές γιατί δεν υπάρχει μια ενιαία κουλτούρα ποινικού δικαίου. Δεν υπάρχει δήμος, παραδείγματος χάρη, για το ε, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Δεν ισχύει το ίδιο Σκανδιναβία, όπου υπάρχει το λεγόμενο σκανδιναβικό ένταλμα σύλληψη και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί ε, και ο λόγος είναι απλούστατος. Στις σκανδιναβικές χώρες ή την Ισλανδία και την Φινλανδία υπάρχει μια κοινή κουλτούρα. Οι νόμοι είναι παρόμοιοι στις χώρες ε, οι γλώσσες επίσης παρόμοιες και κοινέ σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει φόβος ενός, ε, όταν ένας Νορβηγός δικάζεται στη Σουηδία γιατί αντιλαμβάνεται το σύστημα και αντιστρόφως. Αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη, γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε νομίζω να φτιάξουμε ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να οικοδομήσουμε τον Ευρωπαϊκό Δήμο στο θέμα το οποίο ανέπτυξα. Λοιπόν, αυτά αν έχετε ερωτήσεις βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που ήθελα να αναφέρω, αλλά θα τα αφήσω στην οθόνη για να τα διαβάσετε με την ησυχία σας και νομίζω πως ε, έμεινα εντός του χρόνου που ορίσατε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ εμείς. Στη διάρκεια της παρουσίασής σας αναφερθήκατε σε μία σειρά από δυσλειτουργίες οι οποίες ε, νομίζω ότι θα συζητηθούν και τώρα. Να δώσω αμέσω ε, το λόγο στον συγκεκριτή τον κύριο Ιακολίνο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αδιαμφισβήτητα το ποινικό δίκαιο, όπως ε, αναφέρθηκε, ουσιαστικά βασίζεται στην εμπειρία του κάθε κράτους μέλους. Δεν υπάρχει ένα νομικό μοντέλο το οποίο να αφορά όλες τις ε, δικαιοδοσίες. Και στο ποινικό δίκαιο προσαρμοζόμαστε στην κάθε χώρα. Η παράδοση της κάθε χώρας δεν μπορεί να θεωρηθεί ευρωπαϊκή, αλλά είναι εθνική. Το τελευταίο τμήμα της παρέμβασης του δεύτερου μολυτή Ακούσαμε το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ε, το θέμα αυτό ενδιαφέρει όλους μας, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει σχετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δούμε εάν θα παρουσιαστεί, να δούμε αν θα καταφέρει να συγκεράσει τις καλύτερες εμπειρίες, να δούμε αν θα καταφέρει να εγγυηθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όταν υπάρχουν αδικήματα τα οποία ε, περιλαμβάνουν δράστες ή και χαρακτηριστικά σε διάφορες χώρες μέλη. Θα ήθελα να θέσω την εξής ερώτηση εν είδη προβληματισμού. θεωρείτε ότι είναι περίπλοκο ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων, ιδίω των προσωπικών δικαιωμάτων και της προστασία του όταν πρόκειται για αδικήματα τα οποία ε, δημιουργούν ε, ε, κοινωνικό πρόβλημα και ανισορροπία σε κοινωνικό επίπεδο. Το σημείο ισορροπία δεν είναι πάντα εύκολο να το βρούμε και θα δούμε, εάν υπάρξει και Ευρωπαίος εισαγγελέα, τι δυνατότητες έρευνας θα έχει, ε, και κατά πόσον θα ε, μπορέσει να εξισορροπήσει κάποιες καταστάσεις οι οποίες ε, αυτή τη στιγμή είναι εκ διαμέτρου αντίθετες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα σημείο ισορροπίας. Τα εγκλήματα, στο οργανωμένο έγκλημα, στην ομοιοποίηση παρανόμενων εσόδων, στη διαφθορά έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο το γεγονός ότι είναι πολύ σοβαρά αδικήματα και εκεί η προστασία της, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάποιο βαθμό θα πρέπει ε, να ε, υποχωρεί στην αναζήτηση της δικαιοσύνη και στην αναζήτηση ενός τρόπου να επιβάλλουμε δικαιοσύνη. Ευχαριστώ ο κύριος Νιωτοντάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και όσοι είμαστε παρόντες ε, είμαστε πολύ τυχεροί που τι ακούσαμε και λυπάμαι που δεν έχει εδώ άλλου συναδέλφου. Κυρία Κουάσνη, έχω μια σειρά από ερωτήσει. Μια γενική ερώτηση, διότι κατάγομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και τίθεται πάντα. Γίνονται γενικώ κινήσεις για να τροποποιήσουμε τη σύμβαση. Έχουμε 46 μέλη, τώρα ακόμα περισσότερα. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να τροποποιηθεί. Αναφερθήκατε στην ε, συμβατότητα με τις Βρυξέλλες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς όμως έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις οδηγίες και την ομοθεσία και μου φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο στο Συμβούλιο της Ευρώπης να αλλάξει πράγματα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε σχεδόν τίποτα. Έχετε την αρχική σύμβαση από το 1950. Ε, επικρίνεται πολύ στη χώρα μου ακριβώς γιατί δεν μπορεί να αλλάξει και δίνει κάποιες ερμηνείες οι οποίες δεν έχουν πλέον σχέση με τα όσα συνέβαιναν πριν από 60 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να την αλλάξετε. Και δεύτερη ερώτηση. Ένας Βέλγος αστυνομικός πριν από τα Χριστούγεννα μου είπε ότι εργαζόταν στο διαδίκτυο ε, διερευνώντας ε, μία συμμορία οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιείται διαρασυνοριακά και διαπίστωσε ότι του σταμάτησαν τις έρευνες διότι τα ατομικά δικαιώματα ενός από τους δράστες προστατεύονταν από ε, την προστασία των προσωπικών του δικαιωμάτων και αν συνέχιζε την έρευνά του θα παρανομούσε. Και είπε ότι αυτό είναι παράλογο. Έχει δίκιο. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αν δεν μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα η σύμβαση, ε, θα υποχρεωθούμε να σταματήσουμε τα πράγματα. Ε, εγώ δεν είμαι νομικός και θα σας ήμουν ευγνώμων αν ρίξετε λίγο φως σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και μία ακόμα ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια τρίτη. Από ό,τι κατάλαβα, ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων είναι διαφορετικός σε κάθε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι αποδεκτό αυτό και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, διότι δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, διότι κάποιοι εγκληματίες λένε ότι θα φροντίσω να χρησιμοποιήσω ε, ο χρόνο που είναι πιο επιφελής για μένα και θα χρησιμοποιήσω την τάδε χώρα πούμε, που έχει μικρότερο χρόνο διατήρησης και αυτό φυσικά μας δημιουργεί προβλήματα. Και στον κύριο Κρόσμπι τώρα. Ως επιστήμονας, εμένα πάντα με γοητεύουν οι ευφυείς ε, νομικοί, διότι ε, οι περισσότεροι επιστήμονες είναι... Ε, στα όρια της παράνοιας. Δεν τα κατάλαβα όλα όσα είπατε, αλλά πραγματικά με εγωίτευσαν ιδιαίτερα. Αναφερθήκατε στο JD και είπατε ότι οι Αμερικανοί δεν ήταν διατεθειμένοι να τον εκδώσουν. Αυτό είναι παράλογο. Υπάρχει έλλειψη συνεργασίας διότι εμεί θέλουμε να στείλουμε την προσωπία στη Washington τον Απρίλιο και πραγματικά αυτό θα ήταν από τα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μαζί του. Έχω σημειώσει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που είπατε. Θα σταματήσω τώρα και θα ήθελα να επανέλθω όταν καταλάβω τι έχω σημειώσει εδώ, αν μου επιτρέψετε να δευτερολογήσω. Και ελπίζω να μας δώσετε και την παρουσίασή σας με διαφάνειες για να μπορέσουμε να την μελετήσουμε και αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπιλ. Ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Αναφερθήκατε επανειλημμένως στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μετά στην παρέμβασή σας μας δείξατε ότι υπάρχουν μια σειρά αποχάσματα. Αβυσαλέα τα κενά ανάμεσα στην νομοθεσία των κρατών μελών. Molto strana, come in Υπάρχουν τα εξή παράδοξα στην ομολογία κάποιων χωρών δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ενάγοντος ή ορισμένες φορές ε, ε, χρησιμοποιείται ως κατήγορος για να υπάρχει και μεγαλύτερη αντίθεση, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες θεωρείται ότι η εσείς επίσης αναφερθήκατε και στο ρόλο της Eurojust. Ε, εμείς ε, αντιλαμβανόμαστε ότι ορισμένες φορές δεν χρησιμοποιείται η Eurojust από τα κράτη-μέλη, ενώ θα έπρεπε, και ορισμένες φορές ε, την υπερβαίνουν επειδή διάφοροι δικαστές γνωρίζονται απευθείας και διευκολύνονται έτσι καλύτερα, θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να παρέμβει Eurojust. Όταν αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, τι είναι αυτό το οποίο τους ενώνει. Διότι εσείς είπατε ότι για να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτά τα προβλήματα και να είναι ο κατήγορος ακόμα πιο ισχυρός, ε, ο Ευρωπαίος εισαγγελέα και ε, μια ενιαία ε, νομοθεσία θα μπορούσε να διευκολύνει όλες αυτές τις πτυχές. Εμείς βέβαια συνειδητοποιούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να εναρμονιστούν όλα τα ποινικά συστήματα, τα δικαστικά συγγνώμη συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε 27, ε, σχεδόν 28 πλέον διαφορετικοί τρόποι ερμηνεία, ε, για παράδειγμα του οργανωμένου εγκλήματος, διαφορετικές ευαισθησίες από πλευράς ε, δικαστικών, και 27 διαφορετικοί τρόποι αντίληψη του όλου ζητήματος. Στην Ιταλία το οργανωμένο έγκλημα έχει συγκεκριμένη σημασία. Για κάποιες άλλες χώρες, ε, για παράδειγμα εμείς ε, προσπαθήσαμε να δούμε πώς αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, το θέμα αυτό και τι αίσθηση έχουν και πώς θεωρούν ότι είναι το οργανωμένο έγκλημα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι πολίτες θεωρούν ότι οργανωμένο έγκλημα είναι ο αυξημένο αριθμός κλοπή ποδηλάτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τελείω διαφορετικό ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα θέματα σε 27 διαφορετικοί τρόποι. Ε, πέραν του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να διευκολύνουν τα κράτη-μέλη αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο ω προ την εναρμόνιση, αλλά και προ μια ενιαία νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επαναλαμβάνω ότι εγώ είμαι βέβαιη ότι μπορεί να ενισχύσει τις κατηγορίες και μπορεί να αποτελέσει και εγγύηση για τον κατηγορούμενο. Παρακαλώ. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Κουάσνη. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νεύτον Αντάν, για το ερώτημά σας το πρώτο για τις τροποποιήσεις εξυγχρονισμού. Εγώ μιλούσα όχι για τροποποιήσεις της Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά για τις τροποποιήσεις που εξεργαζόμαστε για την ε, οδηγία για τη Σύμβαση Προστασίας των Δεδομένων. Γιατί θέλουμε να παραμείνουμε συμβατοί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο. Δεν αφορά λοιπόν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 47 συμβαλόμενοι ασχολούνται. Αυτή τη στιγμή γίνεται ακόμα η ανάλυση, ξέρω ότι και στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδιαφέρονται, και το κυριότερο θέμα είναι κατά πόσον θα γίνει πανενοσιακό κείμενο. Δεν υπάρχει άλλη τροποποίηση για τον εξυγχρονισμό. Για τη Σύμβαση Προστασίας των Δεδομένων πάντων μιλούσα. Τώρα για το παράδειγμά σας του Βέλγου αστυνομικού Αυτά είπε και ο κύριος Γιακολίνος. Πρέπει να εξισορροπήσουμε την καταπολέμηση του εγκλήματος με την, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν υπάρχουν ύποπτοι ή κατηγορούμενοι κτλ. Είναι δύσκολο πράγμα, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει η Ευρωδίκ και η Ευρωάστε στην Ένωση. Και αυτό επιτρέπει τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και τα εθνικά τι αυτά και άρα δεν είναι ο στόχος μας μη ρεαλιστικός, ουτοπικός γιατί ζητούμε απλώς εναρμόνιση της υπάρχουσας νομοθεσίας που θα διευκολύνει τη συνεργασία. Ε? Συνήθως έχουμε το πρόβλημα πώς να συνδυάσουμε τους διάφορους τομείς και θέματα γιατί η προστασία των δεδομένων αφορά ολόκληρη την κοινωνία και όταν βλέπουμε πράγματα όπως το κυβερνοέγκλημα ή ε, καταλαβαίνουμε ότι πάντα γίνονται τα ίδια σχόλια, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να τα συνδυάσουμε για να καταλάβουν οι διοκτικές αρχές ότι δεν είναι εξτρεμιστικό να ζητάμε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί να επιβληθεί ο νόμος και από αστυνομικούς με το σεβασμό απλών αρχών προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων. Δεν είναι τίποτα παράλογο ή υπερβολικό. Όσο για την παρακράτηση, κατακράτηση, διατήρηση, αποθήκευση δεδομένων, το λέμε και αυτό, το λέμε. Το λέμε. Ε, στα κράτη-μέλη της Ένωσης υπάρχουν διαφορές, αλλά ειδικά για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών υπάρχει κείμενο και προβλέπεται ανώτατη περίοδος κατακράτησης των δεδομένων. Σε μερικές χώρες μέλη όμως επικρίθηκε και αυτό το κείμενο και οι συνταγματικά δικαστήρια το καταψήφισαν, το καταδίκασαν και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Κρόσμπη για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω με τη Eurojust. Έχω την υποψία ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εθνικοί συγγελείς, οι ανακριτές και οι δικαστές τείνουν να μην ε, παραπέμπονται στη Eurojust επειδή δεν γνωρίζουν πολύ καλά τις διαδικασίες, ε, θεωρούν ότι είναι πολύ γραφειοκρατικό, είναι μεγάλο το άχθος και όπως λέτε και στα Ιταλικά ε, να προσπαθούν να μπουν στο προκείμενο, δηλαδή να εξετάζουν το ζήτημα όπως το βλέπουν χωρίς παρεμβολές από άλλους. Ε, υποψιάζομαι λοιπόν ότι δεν χρησιμοποιούμε, δεν εκμεταλλευόμαστε επαρκώς τις δυνατότητες της Eurojust. Αν την χρησιμοποιούσαμε μπορούν να ε, υπήρχε και διευκόλυνση. Τώρα, το θέμα του ενάγοντος είναι ευαίσθητο ζήτημα σε χονδρικές εκτιμήσεις, τώρα το σκέφτηκα αυτό, χονδρικά λοιπόν η μισή Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σύστημα βάσει του οποίου τα θύματα μπορούν να εμφανιστούν στο δικαστήριο στο πλευρό του εισαγγελέα και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Αυτοί που δεν χρησιμοποιούν λοιπόν τη δυνατότητα της μήνυσης και του ενάγοντος ως δεύτερο εισαγγελέα, ως δεύτερο κατήγορο, μπορεί με την παρουσία του μάρτυρα να επιβραδύνουν τη διαδικασία. Να σας δώσω ένα φθαίρετα παράδειγμα. Αν δείτε την υπόθεση με το κρουαζιερόπλιο Κώστα ε, που είχαμε τον περασμένο Ιανουάριο, ε, αυτή η υπόθεση είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια στην Ιταλία και έχουμε 1.500 ε, ενάγοντες, 1.500 θύματα περίπου που συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία κατά του καπετάνιου του σκάφου. Όλου αυτού του ανθρώπου πρέπει να του ακούσουμε και ο καθένα από αυτού θα έχει μια διαφορετική απέτηση. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η δίκη δεν το γνωρίζω, φαντάζομαι χρόνια και οι δίκες στην Ιταλία κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουν. Και το πρόβλημα είναι, ε, αν δεν κάνω λάθος, 10 χρόνια είναι η μέγιστη διάρκεια μιας δίκης και το θέμα είναι ότι μπορεί να παραγραφεί στη συνέχεια, να περάσει ο χρόνος της. Αυτή είναι η δυσκολία. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση βέβαια σε αυτή την περίπτωση. Σε κάποιο βαθμό όμως ε, παραβιάζει τη δυνατότητα της ε, υπεράσπισης. Τι γίνεται τώρα με τις 27 διαφορετικές πραγματικότητες. of course not possible, uh, to... Σαφώς ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εναρμονίσουμε 27 διαφορετικά ποινικά συστήματα. Ακόμα και μεταξύ Σκοτίας και Αγγλίας έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα, τα οποία συμπίπτουν στο πλαίσιο του ίδιου κράτους, ε, τη Μεγάλη Βρετανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο αν θέλετε, αλλά δεν έχουν εναρμονιστεί τα ποινικά του συστήματα και υπάρχει διαφορετικό ανώτατο δικαστήριο για τον καθένα από τους δύο. Ε, Φανταστείτε δεν να το προβάλλουμε αυτό σε μεγαλύτερη κλίμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 κράτη-μέλη και 28, μάλλον είναι δύσκολο. Ή τουλάχιστον δεν είναι εύκολο στο εγγύς μέλλον, ούτε στο μεσοπρόθεσμο μέλλον και σίγουρα δεν θα συμβεί όσο ζω εγώ ε, ή μάλλον όσο ζει ο καθένας από εμά ε, σε αυτή την αίθουσα. Είναι πολύ μακροπρόθεσμο όραμα αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο δημιουργούμε συνεχώς, ελπίζουμε ότι θα διαρκέσει στο Δινεκές και δημιουργούμε κάτι μόνιμο. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποια μέλη που γίνονται πιο δύσκολα και δεν ε, αντιλαμβάνονται μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και δεν έχουν αυτό το όραμα. Πέραν αυτόν όμως κάτι πρέπει να γίνει. Η εναρμάνωση αυτή καθεαυτή θα είναι πολύ σύνθετη. Και ίσως είναι λίγο απλοϊκό αυτό που σας λέω, αλλά θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ένας Ευρωπαίος ε, εισαγγελέα, διότι θα ε, εναρμονίζει σταδιακά. Ο εισαγγελέα θα ξεκινήσει, για παράδειγμα, με εγκλήματα ε, Απάτη, για παράδειγμα, στο κοινοτικό προπολογισμό. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταρτίζεται αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω ότι σε αυτό θα περιοριστεί. Αυτή τη στιγμή ε, δεν νομίζω ότι θα περάσει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πέραν τη προστασία του ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Εάν λοιπόν ε, περάσει όμω αυτό το νομοθετικό κείμενο και έχουμε έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα γι' αυτό, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να διαβρύνουμε τα καθήκοντά του. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ή μάλλον δύο. Αφενός, έχουμε ένα ευρωπαϊκό κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κάποια ε, στοιχεία. Αναφέρομαι στον, ε, στους νόμους περί ανταγωνισμού. Όταν ξεκίνησα εγώ ήταν τα άρθρα 85 και 86 της συνθήκης, ενώ τώρα είναι τα 101 και 102 της συνθήκης. Ήταν ουσιαστικά ευρωπαϊκό δίκαιο. Και η ευρωπαϊκή αυτή νομοθεσία εχωρήθηκε στα κράτη-μέλη μέσω των κανόνων του ανταγωνισμού. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού είναι πλέον ε, σε κυρίαρχο βαθμό ε, δικαιοδοσία των κρατών μελών ε, υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ε, ο νόμος περί ανταγωνισμού ασχολείται με καρτέλ που κανονίζουν τις τιμές, ε, κανονίζουν τα θέματα της παραγωγής και το καθεξής, οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τις αρχές, είτε είναι οι ευρωπαϊκές αρχές είτε είναι οι εθνικές αρχές, βάσει του Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ποινικά αδικήματα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ πιο αυστηροί διαδικαστικοί κανόνες. Και αυτό επιβεβαιώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην περίπτωση Μεναρίνη που είναι μια Ιταλική υπόθεση. Στην υπόθεση Μεναρίνη το δικαστήριο είπε ότι οι κυρώσει είναι ποινική φύσεως και επομένως ε, θα πρέπει να υπάρχουν ενισχυμένα δικαιώματα για την υπεράσπιση. Και σημαίνει επίσης όμως ότι στην ουσία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρεί ότι οι κυρώσει που επιβάλλονται στα καρτέλ είναι ποινική φύσεως. Και αυτό είναι ένα δικαστήριο το οποίο έχουμε επιβάλει εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να γίνει λοιπόν, ναι μεν σε περιορισμένο αλλά, επίπεδο, αλλά βαθμιδών θα φτάσουμε στο σύνολο. Και κάτι ακόμα. Στην Ελβετία, δεν ξέρω πόσα καντόνια έχουμε, αν ξέρει κανείς να μου πει, 20 και κάτι καντόνια, ορίστε. Μέχρι πριν από 100 περίπου χρόνια, κάθε καντόνι στην Ελβετία είχε διαφορετικό ποινικό δίκαιο. Και πολύ συχνά, μεταξύ δύο καντονιών, ε, το ποινικό δίκαιο στο κάθε καντόνι ε, έλεγε εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα. Ε, κάτι το οποίο λοιπόν θεωρείται έγκλημα στο Τούιχ δεν είναι έγκλημα στο Τιτζίνο ή Τούμπαλιν. Και αυτό φυσικά ε, σήμαινε ότι δεν ήταν αποτελεσματική δικαιοσύνη, δεν μπορούσε να υπάρχει συνοχή στην ελβετική ε, κοινωνία και δεν υπήρχε συνοχή στο ελβετικό κράτος. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι κάθε καντόνι ήθελε να διατηρήσει την κυριαρχία του στα θέματα ποινικού δικαίου και επομένως δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στην εναρμόνιση. Και τι έγινε, η Ελβετία επέβαλε ένα κώδικα έναν ελβετικό ομοσπονδιακό ποινικό κώδικα, ο οποίος είναι ακόμα ενισχύ. Η Ελβετία είναι λίγο μικρότερη βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τη χρησιμοποιώ ω παράδειγμα. Αν τα καταφέρνει η Ελβετία, ε, τελικώ θα τα καταφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πρέπει να γίνει στην αρχή στη βάση της ενισχυμένης συνεργασία. Κάποια κράτη-μέλη μπορεί να το επιθυμούν, κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά επειδή κάποιοι δεν το επιθυμούν, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποτελέσει αυτό ανάχωμα στην πρόοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κρόσμπι. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, ο κύριος Σταβάρης θέλει το λόγο. Okay, uh, all, I... Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήμουν στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπότε δεν άκουσα την παρουσίαση ολόκληρη. Αυτό το οποίο έπιασα όμως ήταν ήδη ενδιαφέρον. Και έχω κάποια πράγματα που θα ήθελα να πω. Χτες συζητήσαμε πολύ το... Αυτό το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα ειδικά τους φιλελεύθερους, ένα ε, ευρωπαϊκό FBI. Που πάει ακόμη παραπέρα από αυτό το οποίο προτείνεται. Στις είπα πρόκειψε κάπως αργά, ε, από ό,τι θυμάμαι στην ιστορία της χώρας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κάτι, εάν δεν είπατε κάτι στη διάρκεια της παρουσίασης. Επίσης, αν ε, έχετε κάποιες σκέψεις για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαίου Εισαγγελέα και Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εάν η εισαγγελέα ξεκινήσει μόνο με την δίωξη εγκλημάτων εις βάρος του ευρωπαϊκού προπολογισμού, αλλά τι θα γίνει με την προληπτική δίωξη δικημάτων ή τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, και λόγω της ιστορικής εμπειρίας της ε, Ελβετίας και άλλων συνομοσπονδιών, ε, δημοκρατικών πολιτιών γενικώ. Ποια στοιχεία θεωρείται ότι θα ήταν τα πρώτα στοιχεία ενός ε, ευρωπαϊκού πλαισίου. Έχετε το λόγο. Πριν απαντήσω, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Νιούτον Τάν γιατί δεν απάντησα για την έκδοση από τη ΣΥΠΑ. Κοιτάξτε, όσον αφορά την έκδοση, η κλασική θέση των περισσότερων κρατών είναι πως δεν εκδίδουν ε, υπηκόους τους. Εκτός εάν ε, υπάρχουν σοβαροί λόγοι. να σας δώσω και ένα άλλο αυθαίρετο παράδειγμα. Υπάρχει συνθήκη έκδοσης ε, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη, το Ηνωμένο Βασίλειο θα ε, εκδώσει τους, ε, θα εκδίδει τους πολίτες του χωρίς δεύτερη σκέψη, ε, ενώ δεν κάνει το ίδιο είπα. Ε, φοβερή ανισορροπία. Και ο λίγος είναι πως στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχουν συνταγματικές δικλείδες ασφαλής γιατί δεν υπάρχει σύνταγμα που θα κατοχυρώνει κάτι τέτοιο. Οπότε είναι ο κατηγορούμενος στο έλεος της πολιτικής διαδικασίας. Οπότε, εν ολίγης, είπα, δεν εκδίδουν τους πολίτες τους. Εκτός εάν είναι θέμα εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Τώρα για να απαντήσω στο δεύτερο κύριο ερωτήσεων. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τις εύκολες. Το πρώτο στρώμο, αν θέλετε, έτσι, κοινών διατάξεων υπάρχει ήδη στην ΕΣΔΑ και στη Χάρτα. Βασικά δικαιώματα όπως ε, το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, το τεκμήριο αθωότητας, ε, το να μην κατηγορείται κανείς ε, δύο φορές για το ίδιο πράγμα. Αυτό το οποίο λέμε στα λατινικά «ne bis in idem». Αυτά τα πράγματα υπάρχουν ήδη σε οριζόντιο, σε πανευρωπαϊκό δηλαδή επίπεδο και θα, θα έπρεπε να γίνονται σεβαστά, δεν γίνονται πάντα και από τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπάρχει ήδη αυτό και μάλιστα το ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, έχουν υπογράψει την ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, ε, επιτρέπει την ανάπτυξη της θεωρίας της αναγνώριση. αναγνώρισης. Δηλαδή όλοι ε, έχουμε κάποιες κοινέ διατάξεις, οπότε οτιδήποτε γίνεται σε κάποιο κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο από όλα τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα είναι η αμοιβαία αναγνώριση. Είναι μια έννοια η οποία δεν έχει σχεδιαστεί για το ποινικό δίκαιο. Αφορούσε την ελευθερία κίνηση αγαθών και υπηρεσιών το Κασίς Dijon, Από εκεί είχε ξεκινήσει. Δηλαδή αν κάτι ε, μπορεί να πωλείται στη Γαλλία, μπορεί να πωλείται και στην Ιταλία. Αυτή είναι η αμοιβαία αναγνώριση. Δεν ε, σημαίνει ότι λειτουργεί αυτομάτως ε, στο, στον ποινικό τομέα. Αλλά υπάρχει λοιπόν ένα πρώτο στρώμα, αν θέλετε, αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχουν ε, διάφορες περιπτώσεις, ανέφερα τον Ebis in Idem, αν ε, υπάρχουν παραδείγματο χάρη ζητήματα προφυλάκησης και της διάρκειάς της. Ε, επίσης ε, υπάρχει η, η εγγύηση με την υποχρέωση μετά να παρακολουθεί το ύποπτος κτλ. λοιπά. Δεν το κάνει αυτό κάθε χώρα. Ειδικά όταν κάποιο είναι υπηκό άλλη χώρα. Γιατί ε, υπάρχει ο φόβο ότι θα φύγουν από τη χώρα και δύσκολα θα ξαναγυρίσουν. Υπάρχει επίση πρόβλημα υπερπληθισμού των φυλακών. Βγήκε μια απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα που καταδίκαζε ένα νότιο κράτος μέλος για απάνθρωποι... Ε, άνθρωπο, επίπεδο υπερπληθυσμού των ε, φυλακών. Και αυτό είναι πρόβλημα για την εκτέλεση ε, των ε, ενταλμάτων σύλληψης. Γιατί ένα κράτος θα το σκεφτεί σοβαρά να στείλει κάποιον σε ένα άλλο που είναι απαράδεκτες συνθήκες στις φυλακές. Και υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Αναφέραμε επίσης το πρόβλημα του ανάγοντος. Πώς λύνεται αυτό. Μπορεί να υπάρξει ένα συμβασμό, δεν ξέρω. Ένα άλλο ζήτημα. Ε, είναι το θέμα των δικών με ενόρκους. Π.χ. στις βαλτικές χώρες θεωρείται κάτι το οποίο δεν βοηθάει, έτσι το λέμε. Σε άλλες χώρες βεβαίως η δίκη από ενόρκους είναι βασικό ζήτημα. Οπότε πώς επιλύονται αυτές οι διαφορές. Και, και άλλα πολλά. Τι θέλω να πω λοιπόν. Είναι μεγάλα προβλήματα αυτά. Και ίσως να μην επιλύονται κιόλα. Αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Δεν λέμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και το αποφεύγω. Όχι κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο λίγο. Για ευρωπαϊκό FBI τώρα. Νομίζω ότι χρειάζεται. Χρειάζεται γιατί σε κάποιες περιπτώσεις οπωσδήποτε δεδομένων των πολιτικών πιέσεων μπορεί να μην ε, υπάρξουν διώξεις ενώ θα έπρεπε. Εάν υπήρχε ένα ευρωπαϊκό FBI και εισαγγελέα με επαρκή εξουσίες ίσως να μην ε, ε, είχε τις ίδιες πιέσεις ο εισαγγελέα για να, για να μην ασκήσει δίωξη. Και έτσι να υπήρχε έτσι κάπως μεγαλύτερη αποτρεπτική ισχύς. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Κουάσνη και τον κύριο Κρόσμπι. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας και για το γεγονό ότι μας παρουσιάσετε τις απόψεις σας. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τους κυρίους Όλιβερ Τέιλ και τον κύριο Μάρτιν Μπόζε να έρθουν εδώ στο Προεδρείο. Θα τους ακούσουμε στο δεύτερο τμήμα στα δικαιώματα υπεράσπισης στις διασυνοριακές έρευνες και την δικαστική συνεργασία. Ο κύριος Τέιλ είναι επικεφαλής ε, στη Γενική Διεύθυνση Justice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα μας μιλήσει για το συντονισμό και το δικαίωμα στην υπεράσπιση, ενώ ο κύριος Μποζέ είναι από το Πανεπιστήμιο της Βόνης και θα μας πει για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και τις επιπτώσεις που έχει στην υπεράσπιση. Και πάλι από 15 λεπτά ο καθένας. Θα ξεκινήσει λοιπόν ε, ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Justice και από εκεί και πέρα θα ακούσουμε τον καθηγητή Μποζέ. Εγώ ζητώ συγγνώμη, θα φύγω εντός λίγο και θα αναλάβει τα ενία της Προεδρίας ο κύριος Ταβάρες. Παρακαλώ. Merci Σας κατευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. καθώς και την Επιτροπή σας ολόκληρη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Ο στόχος της Ένωσης, καλό είναι να το επιθυμίσουμε, είναι να δημιουργήσει ένα πραγματικό χώρο ευρωπαϊκής δικαιοσύνης μέσα στον οποίο οι πολίτες να είναι βέβαιοι ότι τα δικαιώματά τους αναγνωρίζονται και τη χάνουν προστασίας από την ποινική οικονομία όποιος και να είναι ο χώρος όπου βρίσκονται. Σε, δύο, σε τρία τμήματα θα χωρίσω την ομιλία Καταρχήν το ιστορικό. Μετά η σημερινή κατάσταση και ύστερα οι προοπτικές του μέλλοντος. Μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, η πρόοδος της ποινική δικονομίας στην Ευρώπη ήταν περιορισμένη και τονίζαμε κυρίως θέματα ασφαλείας. Στα ποινικά ήταν περιορισμένη η δράση της Ένωσης λόγω των κανόνων που ονομάζονται του τρίτου πυλώνα που απαιτούν ομοφωνία και υπάρχουν πολύ περιορισμένες δικαιοδοσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πριν από τη Λισαβόνα η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφερόταν για την εναρμόνιση του υλικού δικαίου, δηλαδή την ενέκρινε πολλά κείμενα για την ενδυνάμωση της εναρμόνισης των κυρώσεων στα θέματα ξεπλήματος βρωμίκου χρήματος, ε, εμπορία ανθρώπων κλπ. Για τα ποινικά λοιπόν η Ένωση ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την αμοιβαία αναγνώριση των ε, δικαστικών αποφάσεων. και οι συζητήσεις που γίνονταν με πρωτοβουλία της Κομισιόν δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αντίθετα, σημειώθηκαν σημαντικές προόδοι στο θέμα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για να διευκολυνθούν εδιώξεις. Εργαλεία δικαστικής ποινική συνεργασίας έχουν εγκριθεί, το πιο γνωστό είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ώστε όσοι είναι ύποπτοι κάποιου εγκλήματος να μπορούν να δικαστούν παντού στην Ευρώπη. Υπάρχει η Συμφωνία Δικαστικής ε, Συνεργασίας του 2000 για το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων τις κατασχέσεις κλπ. Υπάρχουν λοιπόν εργαλεία συνεργασίας. Και ενδυναμώθηκαν ιδίω με τη δημιουργία και την ενδυνάμωση του 2008 της Eurojust που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μεικτών ομάδων έρευνας και όλα αυτά δείχνουν τις δυνατότητες της Ένωσης να δώσει στους δικαστάς ε, και τους εισαγγελείς εργαλεία συνεργασίας. Αντίθετα, πριν από τη Λισαβόνα λίγα είχαν γίνει για την προστασία των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων και υπόπτων. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επανεξισορρόπηση του συστήματος. Η στρέβλωση που σημειώνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ των δικαιωμάτων της υπεράσπισης στις διάφορες χώρες είναι μια ανομαλία που πρέπει να διορθωθεί. Σας υπενθυμίζω ότι παραδοσιακά συνήθως δηλαδή η ποινική δικονομία στοχεύει στην ταύτιση και τιμωρία των παραβατών και απαιτείται η εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων για τη διαπίστωση κτλ. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται στην καρδιά η ποινική οικονομία των δημοκρατικών εγγύσεων. το δικαίωμα δηλαδή σε μια δίκαιη δίκη. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ αντίφαση μεταξύ δικαστικής συνεργασίας και εγγύησης των ατομικών δικαιωμάτων. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Αυτή η ποινική συνεργασία είναι απαραίτητη. Εδώ είμαστε στην Επιτροπή σα και θα πρέπει να πούμε ότι για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα, χάρη την εμπορία ανθρώπων, την ε, ε, ε, εμπορία ναρκωτικών κλπ., πρέπει να ενδυναμωθεί η συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος και που έχει εξορισμού διεθνικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, η εξισορρόπηση των ποινικών διαδικασιών στις χώρες μέλη περνάει και από την εγγύηση των δικαιωμάτων της υπεράσπισης του κατηγορουμένου ή του υπόπτου που υπενθυμίζω ότι μέχρι την τελική του καταδίκη θεωρείται αθώος. Πρέπει λοιπόν να ενδυναμωθούν όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε και τώρα και στο μέλλον για να υπάρξουν να δοθούν σημαντικές εγγυήσει για τα δικαιώματα των προσώπων. Σήμερα η συνθήκη της Λισαβόνας μας επιτρέπει να εξισορροπήσουμε τη δράση μας και να βασιστούμε στα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη η χάρτα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή από όλους τους πολιτικούς και όλα τα πολιτικά μας προγράμματα. Σήμερα, τώρα, προετοιμάζουμε μία πρόταση για την ενίσχυση όλων αυτών γιατί για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Πρέπει όλοι όσοι είναι, εμπλέκονται σε μια ποινική διαδικασία είτε είναι ύποπτοι είτε είναι θύματα να προστατεύονται όπου και να κατοικούν στην Ένωση. Η πρώτη φάση ήταν η έγκριση της διαδικασίας, της ε, οδηγίας που διασφαλίζει τα δικαιώματα αυτά για όλους τους κατηγορουμένους υπόπτους όταν ας πούμε δεν μιλούν την ίδια γλώσσα με τους δικαστάς και προβλέπεται η μετάφραση και διερμηνία όλων των φάσεων της διαδικασίας. Υπάρχει λοιπόν εδώ θέμα δικαιώματος στην πληροφόρηση ως προς τα δικαιώματα και τις κατηγορίες που έχουν απευθυνθεί και που μέχρι τις 2 Ιουνίου 2014 πρέπει να έχει εγκριθεί και μεταφερθεί Θα υπάρχει δηλαδή ένα έγγραφο που θα χορηγείται σε όλους τους κατηγορουμένους με τα δικαιώματά του, το δικαίωμα να σιωπήσει, να έχει δικηγόρο, να έχει μετάφραση και διερμηνία, ιατρική εξέταση κτλ. Η οδηγία αυτή περιλαμβάνει και διατάξεις για το δικαίωμα πρόσβασης στο ποινικό φάκελο του κατηγορουμένου. Επίσης προτείναμε μία οδηγία για, ειδικά για την πρόσβαση σε δικηγόρο τον Ιούνιο του 2011 και ως προς το δικαίωμα επικοινωνίας με την οικογένεια του κατηγορουμένου ή του υπόπτου. Αυτό είναι ο ακρογωνίος λίθος των προσπαθειών μας γιατί το δικαίωμα στην αρρωγή από δικηγόρο είναι η βάση όλων των υπολείπων δικαιωμάτων. Από την αρχή ήδη της διαδικασίας πρέπει να χορηγείται δικηγόρος γιατί είναι κάτι τελείως απαραίτητο για να υπάρξει δίκαιη δίκη. Αυτά βασίζονται βέβαια στο κεκτημένο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά είναι και ένα γενικότερο αυξημένο επίπεδο προστασίας γενικά στην Ένωση. Τώρα για το μέλλον. Χρειάζεται ακόμα να υπάρξουν και άλλες προσπάθειες για να συμπληρωθούν όλα αυτά. Οι πρωτοβουλίες μας είναι ειδικέ εγγυήσεις για τους υπόπτους ή κατηγορουμένους ιδιαίτερα που βρίσκονται σε λεπτή θέση όπως παιδιά. Μία πρόταση πρωτοβουλία για την δικαστική αρρωγή για τους υπόπτους ή κατηγορουμένους που είναι και αυτό σημαντικό για να εφαρμοστεί το δικαίωμα της πρόσβασης σε δικηγόρο για όποιον δεν έχει πόρους για να πάρει δικό του δικηγόρο και όπως είπε και η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ μια άλλη πρωτοβουλία για να ενισχυθεί το δικαίωμα του υπόπτου σε αθωότητα μέχρι να καταδικαστεί. Σας υπενθυμίσω ότι τον Ιούνιο του 2011 επίσης η Κομισιόν υπέβαλε μια πράσινη βίβλο για την κράτηση για όλες τις, τις φάσεις και που τονίζει ιδιαίτερα το θέμα της προφυλάκησης. Υπερβολικά μακρές περίοδοι προφυλάκησης ή η συστηματική της χρησιμοποίηση, ιδίως από ξένους, είναι κάτι που μπορεί να υπονομεύσει την δικαστική συνεργασία και δεν ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές της Ένωσης. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ενδυναμώσουμε τη μεταφορά όλων αυτών στα εθνικά δίκαια ιδιαίτερα ως προς την κράτηση η απόφαση πλαίσιο συγκεκριμένα για τα μέτρα επιτήρησης European Supervision Order το λέμε για να διευκολυνθεί έτσι η εξέβρεση εναλλακτικών λύσεων προς την προφυλάκηση. Τέλος, για την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη σημαίνει ότι οι δικαστικές αρχές πρέπει να έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη κατά την εφαρμογή των αρχών της ισονομίας και δικαιοσύνης και σημαίνει επίσης ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην, στον δίκαιο χαρακτήρα των διαδικασιών και να είναι σίγουροι ότι θα τύχουν σεβασμού των δικαιωμάτων τους όποτε κατηγορούνται σε κάποιο δικαστήριο που δεν είναι της χώρας τους. Αυτό φυσικά αφορά την ποιότητα της δικαιοσύνης και όπως το υπενθύμησε επίσης η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ, οποιοδήποτε κυκλοφορεί στην Ένωση πρέπει να μπορεί να αναμένει ότι παντού θα βρει μια δικαιοσύνη υψηλού επίπεδου. Είναι κάτι που το ζητούν και όλοι οι πολίτες. Αλλά για να λειτουργήσει αυτό βέβαια πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αυτή την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να ενδυναμωθούν τα δικαιώματα. Η εναρμόνιση των κανόνων της δικονομία θα ενδυναμώσει και την εμπιστοσύνη των κρατών μελών στα δικά τους ε, δικαστικά συστήματα καθώς και των υπολείπων χρόνων. Σας κατευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε για αυτά που είπατε και δίνω το λόγο τώρα στον καθηγητή Μπόζερ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για να μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, και την επίδρασή του στα δικαιώματα της υπεράσπισης. Ε, πρέπει να ξέρουμε καταρχήν για να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση το status quo ante το προηγούμενο καθεστώς. Βεβαίως ε, έχουν αλλάξει ριζικά τα πράγματα με το νέο αυτό μέσω το Ευρωπαϊκό Εντάλμα Σύλληψης. Αλλά θα δείτε πως περισσότεροι από αυτούς τους κανόνες που αναφέρονται στην απόφαση πλαίσιο ε, υπάρχουν ήδη στους κλασικούς κανόνες έκδοσης ε, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοση 1957, την ε, Συμφωνία Σέγγεν και την ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση 1996 για την έκδοση. Ποια είναι τα καινούργια πράγματα λοιπόν. Μία σοβαρή αλλαγή είναι πως έχουμε μια γρήγορη διαδικασία. Υπάρχουν αυστηρές προθεσμίες για την έκδοση και έχουμε τώρα απλά τις ε, έχουμε δίκες μόνο για τις περιπτώσεις έκδοσης οπότε έχουμε κάποιες ε, παραδοσιακές διαδικασίες δεύτερον έχουν καταργηθεί κάποια παραδοσιακά εμπόδια που υπήρχαν δηλαδή το διπλό αξιόπινο το ότι δεν εκδίδονταν υπήκοοι και βεβαίως το ότι δεν υπήρχαν εκδόσεις για πολιτικά ε, δημοσιονομικά και στρατιωτικά δικήματα. Οπότε πώς επηρεάζονται έτσι τα δικαιώματα της υπεράσπισης. Α, εφόσον το Ευρωπαϊκό Τέλμα Σύλληψη είναι ένα μέσο για την ε, παράδοση υπόπτου ή καταδικασμένου ανθρώπου δεν ασχολείται με τα δικαιώματα της υπεράσπισης στην ε, ποινική δικονομία στο κράτος μέλος που εκδίδει, αλλά ασχολείται μόνο με την διαδικασία της έκδοσης. Και εδώ πέρα υπάρχουν κάποια βασικά δικονομικά δικαιώματα που ορίζονται στην απόφαση πλαίσιο, όπως το δικαίωμα παρουσίας ε, δικηγόρου και διερμηνέα αν αυτό χρειάζεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και το ε, δικαίωμα μιας ακρόασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14. Αυτό είναι κάτι το καινούριο όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνθήκες και την παραδοσιακή διαδικασία έκδοσης, αλλά όλα αυτά είναι σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους που εκτελεί την έκθεση. Οπότε έχουν ακόμα κάποια διακριτική ευχαίρεια τα κράτη-μέλη όταν μεταφέρουν την ε, νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο και άρα έτσι μπορεί να γίνουν και αναποτελεσματικά αυτά τα δικαιώματα. Παραδείγματο χάρη η ε, αποτελεσματική υπεράσπιση στις ε, περιπτώσεις αυτές εξαρτώνται από το καθεστώς ε, νομικής βοήθειας, δηλαδή το εάν είναι υποχρεωτική η παρουσία δικηγόρου ή όχι και βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και περιορισμοί όσον αφορά το δικαίωμα της τυχόν ακρόαση. Παραδείγματος χάρη στην Γερμανία κάτι τέτοιο είναι μάλλον η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Επιπλέον τα ατομικά δικαιώματα μπορούν να θεωρηθούν ως λόγος απόρριψης του αιτήματο στα άρθρα, όπως αναφέρουν στα άρθρα 3, 4 και 5 και το κράτος το οποίο εκτελεί το ένταλμα, παραδείγματο χάρη, μπορεί να αρνηθεί εάν έχει υπάρξει μία καταδίκη ερήμην καθώς ε, μπορεί να θεωρήσει πως ε, έχει δικαίωμα καταδικαστεί σε μία νέα δίκη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4. Βεβαίως οι περισσότερες ε, από, αυτές, από αυτούς τους λόγους για να αρνηθεί ένα κράτος να εκτελέσει το ένταλμα δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι μια επιλογή του κράτους μόλις και άρα έχει έτσι την διακριτική ευχαίρεια να επιλέξει αν θα εκτελέσει το ένταλμα ή όχι. Οπότε θα λέγαμε πως ε, οι διασφαλίσεις αυτές ε, είναι κάπως ασθενείς και ειδικά όσον αφορά την ε, καταδίκη ερήμην υπάρχει και κάτι άλλο στην απόφαση πλαίσια κλίν και από κάποια σημεία του συνταγματικού δικαίου κάτι το οποίο έχει συζητηθεί στην περίπτωση Μαλώνη όπου ο ύποπτος ε, διέφυγε και ε, μετά ζητήθηκε από την Ιταλία η έκδοσή του για να εκτελεστεί η ποινή που του επιβλήθηκε η Ρήμιν και θεωρείται πως αν δεν εμφανίστηκε στη δίκη δεν άσκησε το δικαίωμά του να είναι παρόν σε αυτήν. Εάν όμως κατηγορείται για κάτι το σοβαρό, βεβαίως ε, αυτό δεν ισχύει γιατί δεν εμφανίζεται στο δικαστήριο απλά γιατί φοβάται ε, ότι θα συλληφθεί. Σύμφωνα με το Εθνικό Δικαίωμα στα περισσότερα η γενική αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα που συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 1 παραγραφος 3 της απόφασης πλαισίου ε, προβλέπει κάποιον επιπρόσθετο και υποχρεωτικό λόγο για άρνηση εκτέλεσης. Μπορεί λοιπόν τα κράτη-μέλη να αρνηθούν να εκτελέσουν ευρωπαϊκό ένταλμα μόνο εάν εκπληρώνονται οι όροι για μια τέτοια αρνητή αιτία. Στην ε, περίπτωση λοιπόν ε, Ράντου, ο Γενικό Εισαγγελέα Σάρπστον στην αιτιολόγηση τη ε, απόφαση είπε πω σε εξαιρετικέ περιπτώσει το κράτο το οποίο οφείλει να εκτελέσει το ένταλμα μπορεί να αρνηθεί να εκδώσει ένα άτομο εάν έχουν παραβιαστεί ή θα παραβιαστούν τα δικαιώματά του αν ακολουθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες κράτησης ε, ε, δεν είναι αυτές τις οποίες ορίζει το άρθρο 3 της ε, ΕΣΔΑ. Ένα άλλο θέμα το οποίο τίθεται είναι και το ζήτημα της αναλογικότητας. Εάν ε, εκδοθεί για πτέσματα ευρωπαϊκό ε, ένα τέτοιο ευρωπαϊκό τέλμα σύλληψης θα πρέπει να μην εκτελεστεί γιατί είναι δυσανάλογο. Συνοψίζοντας ο οι ρυθμιστικές επιπτώσεις που έχει στα δικαιώματα της υπεράσπισης ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι περιορισμένες. Η απόφαση πλαίσιο περιορίζει τις δυνατότητες των κρατών να αρνηθούν να προχωρήσουν σε έκδοση και δεν απαιτεί ε, από τα κράτη-μέλη μέχρι στιγμής να αλλάξουν την ε, σχετική της νομοθεσία. Όμως, η αποτελεσματικότητα του νέου μέσου έχει μια ε, πραγματική επίδραση στην άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Όπως είπα, έχουμε τώρα μια διαδικασία γρήγορη. Η μέση διάρκεια των διαδικασιών υπό το παλιό καθεστώς ήταν γύρω στους 9 μήνες και τώρα είναι γύρω στους 50 μέρες. Και όσο πιο αποτελεσματικές γίνονται αυτές οι διαδικασίες, τόσο πιο αποτελεσματική πρέπει να είναι και η υπεράσπιση. Αυτό οφείλεται και στην αρχή των, των ε, ίσων δυνάμεων που πρέπει να υφίσταται. Και βεβαίως θα πρέπει να ισχύει και η αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και όσο πιο αποτελεσματικό είναι το διεθνέ δίκαιο σε αυτή την περίπτωση, τόσο πιο αποτελεσματική πρέπει να είναι και η υπεράσπιση. Παραδείγματο χάρη, αν δεν μπορεί να παρουσιάσει κάποια αθωωτικά στοιχεία στο κράτο το οποίο εκτελεί την έκδοση, θα πρέπει να έχει δυνατότητα να τα παρουσιάσει στο κράτο το οποίο έχει ζητήσει την έκδοση. Εν ευθέτω χρόνο. Και εδώ πέρα ακριβώ τίθεται το ζήτημα τη ε, εκπροσώπηση. Δηλαδή, η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνο στο κράτος το οποίο κάνει την έκδοση, αλλά και το κράτο το οποίο εκδίδεται κάποιος για να υπάρχει ακριβώς αυτή η διεθνής υπεράσπιση. Και αυτό είναι ε, ουσιαστικό για την υπεράσπιση του συλληφθέντο και για την κατάληξη της ε, υπόθεσης ε, και στα δύο κράτη, ειδικά όταν μιλάμε, όπω είπα, για πτέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσουμε το λόγο για ερωτήσει. Ξεκινάμε με τον κύριο Ιακολίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τους ομιλητές μας για τις ε, παρεμβάσεις τους που είναι πολύ αξιόλογες. Για την πρώτη παρουσίαση λοιπόν του κυρίου όσον αφορά τις ε, προτάσεις που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, καταρχάς για το ότι οποιοδήποτε είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντέου και επίσης ε, για τα θέματα της προσωρινής κράτησης εν ώψη εκδίκασης της υπόθεσης. Υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις, όπως για παράδειγμα και το δικαίωμα του κατηγορούμενου μέχρι να καταδικαστεί Και φυσικά και το θέμα που θίξατε, το γεγονός ότι υπάρχει σύνοστης στα σοφρονητικά καταστήματα, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες, είναι πολύ σημαντικό ποσοστό των κρατουμένων είναι υπήκοοι άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών και στην Ιταλία όπως και στην Ισπανία και στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός ο αριθμός των κρατημένων που είναι ε, υπόδικοι και είναι αναμονή της απόφασης. Και Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέμβουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε αφενός ε, τα δικαιώματα του ατόμου που κατά την άποψή μου είναι αδιαμφισβήτητα και για αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να μας πει και δύο-τρία περισσότερα πράγματα ο κ. Στέλ και να μας πει και τι άποψη έχει επί του ζητήματος ε, και της λεγόμενης ε, σοβαρής κάθερξης που προβλέπεται στην Ιταλική νομοθεσία και χρησιμεύει απλώς ε, ώστε ο καταδικασμένος επικεφαλής της μαφίας που βρίσκεται στη φυλακή να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλους και να δίνει εντολές ε, ακόμα και όταν βρίσκεται στη φυλακή. Ε, είναι μια διαδικασία που μας επιτρέψε να έχουμε σημαντικά στοιχεία και είναι και θέμα ασφαλείας του ατόμου. Θα ήθελα να μας πείτε ένα-δυο πράγματα λοιπόν για το θέμα αυτά και να σας υπενθυμίσω ότι το 2009 με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είχαμε προβλέψει τότε αλλά δεν εφαρμόστηκε τελικώς αυτή η διάταξη και ε, χρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, διέμβρηση ή την ε, ανακαίνιση σοφρονιστικών καταστημάτων που βρίσκονται στην κατάσταση που σας ε, ε, ε, είπα ότι υπάρχει μεγάλη παρουσία κρατουμένων από τρίτες χώρες. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλές οι παρουσιάσεις και ομολογώ δεν τις κατάλαβα. Δεν είμαι νομικός και με ξεπερνούν όλες αυτές οι έννοιες. Μία πολύ απλή ερώτηση στον κύριο Μπόζη για το ένταλμα σύλληψη. Ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ισχύει και για την Νορβηγία και την Ελβετία. Δεν το γνωρίζω και θα ήθελα απλώ να μου απαντήσετε. Και μία ερώτηση προ του δύο. όπω γνωρίζετε, ο στόχο αυτή τη επιτροπή είναι να κάνει μία απόπειρα να ε, δώσει ένα σύνολο συστάσεων προ τα κράτη-μέλη ώστε να κάνουν κάτι για το πρόβλημα του οργανωμένου εγκλήματο. Θα μπορούσατε ίσως να μας δώσετε κάποιες συστάσεις εσείς. Τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να προτείνουμε. Ο εισηγητής ε, συλλέγει στοιχεία ε, για την έκθεση και εμείς συνεισφέρουμε ώστε να προσπαθήσουμε να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει. Τι προτείνετε εσείς. Βέβαια στη συνέχεια θα μπορούμε να τις βελτιώσουμε και να τις τελειοποιήσουμε, αλλά τι θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάποιες ερωτήσεις και θα τις πω στη γλώσσα μου, τα πορτογαλικά. Mm. Σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνετε πορτογαλικά θα σας δώσω λίγο χρόνο για να βάλετε τα ακουστικά σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Τέλ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τι άποψη έχετε για τις διαπραγματεύσεις για το δικαίωμα σε συνήγορο. Πρόκειται για ένα δικαίωμα το οποίο σε κάποια κράτη-μέλη και στο δικό μου είναι αδιαμφισβήτητο. Ένας πολίτης μπορεί να έχει μαζί του συνήγορο, είτε πρόκειται για ποινική διαδικασία είτε όχι, είτε πρόκειται για επαφές με διοικητικές υπηρεσίες και το καθεξής. Το δικαίωμα λοιπόν σε συνήγορο. Ε, για μας είναι ένα πολύ ευρύ θέμα ε, ενώ γνωρίζω ότι κάποιες άλλες χώρες έχουν δισταχμούς επί του θέματος. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε προς τα πάνω αυτή την ε, παρουσία του συνηγόρου, ιδίως όσον αφορά οικονομικά εγκλήματα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας επ' αυτού. Επόμενο ζήτημα. Οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα ποια είναι τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα ε, που προβλέπουν οι συνθήκες Παραδείγματος χάρη το άρθρο 151, το οποίο προβλέπει προηγούμενη διαβούλευση με τα συνδικάτα, οργανώσεις εργαζομένων, σε περίπτωση που υπάρχει ε, συζήτηση περί εργασιακού δικαίου. ή όταν υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις ε, στα εργασιακά δικαιώματα. Είναι λογικό αυτό. Οι πολίτες ε, μπορούν ε, να προσφύγουν στο δικαστήριο για να διασφαλίσουν, για παράδειγμα, ότι θα γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους. Ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 151 εφαρμόζονται όπως πρέπει. Και Μία ερώτηση για την Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει νομοθεσία για το δικαίωμα στην υπεράσπιση ή ε, θα δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές απλώς και μόνον. Ότι εάν δεν υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει περίπτωση να είναι πολύ πιο δύσκολη η ε, πρόσβαση σε δικηγόρο ε, για κάποιον ο οποίος ε, έχει να κάνει με μια διεθνή υπόθεση. Υπάρχουν βέβαια εξειδικευμένοι δικηγόροι που αναλαμβάνουν τέτοιες διεθνείς υποθέσεις, αλλά μπορεί ένας φτωχός πολίτης να έχει πρόσβαση σε τέτοιες μορφής υπεράσπιση. Ε, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει κάτι επιπλέον των κατευθυντηρίων γραμμών επί του ζητήματος. Ναι. Κατόπιν. Πότε έχει πρόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για θέματα προληπτικής κράτησης, εν αναμονή της ε, απόφασης. Τώρα, να περάσω στον κύριο Μποζέ και να συνεχίσω σε αυτά που είπε ο κύριος Νοτοντάν. Εγώ ήμουν εισηγητής για το Κοινοβούλιο για τη συμφωνία έκδοσης ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγίας. Νομίζω ότι είναι καλές οι συνθήκες στι φυλακές της Νορβηγία, Δεν γνωρίζω βέβαια και πολλά. Αλλά είχαμε την τρομοκρατική επίθεση του Μπρέβικ. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τις νορβηγικές αρχές. Υπάρχει και το θέμα της ε, διπλής ποινή και διπλής καταδίκης. Ε, δεν ε, είμαι νομικός. Κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι υπάρχει διπλή καταδίκη. Υπάρχει, για παράδειγμα, το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Αν ένας παράνομος μετανάστης βρίσκεται στη χώρα μου, τι μπορεί να συμβεί σε αυτή την περίπτωση. μου φαίνεται λίγο υπερβολικό να μην μπορεί να εκδοθεί κάποιος για ένα έγκλημα, διότι η μία χώρα μπορεί να θεωρεί ότι είναι πολύ σοβαρό και σε μια άλλη χώρα στο νομικό της σύστημα να θεωρείται ότι δεν αποτελεί έγκλημα το συγκεκριμένο αδίκημα. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι σφάλμα. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την άποψή σας. Και επίσης, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πραγματικά λόγος ε, ε, μεγάλων αποκλήσεων. Είναι απλώς θέμα χρηματοδότησης. Αν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει την κατάλληλη χρηματοδότηση, τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια πράγματα. Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή και ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης περιλαμβάνει αρκετά κενά αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να το επανεξετάσουμε, θα πρέπει να το ε, μεταρρυθμίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις απαντήσεις του κυρίου Τέλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο ερώτημα που μου έθεσε ο κύριος Ιακολίνο για το θέμα της ε, κράτησης, κυρίως της προσωρινής κράτησης. Αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το εξής. Υπάρχουν ε, μέσα που αφορούν την προσωρινή κράτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στόχο έχουν να μειώσουν ε, τη χρήση αυτής της προσωρινής κράτησης και να χρησιμοποιούνται εναλλακτικέ λύσεις από, ε, σε περίπτωση φυλάκισης τα κράτη-μέλη τη μεταφέρουν και θα πρέπει να τις εφαρμόσουν. Έχει καθυστερήσει το θέμα της ε, μεταφοράς ε, για τους κρατουμένους και το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης ε, των αποφάσεων της αποφυλάξης υπό όρους. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Εποπτείας, European Supervision Έντος, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή. Ε, αυτή τη στιγμή τα μισά έχουν μεταφέρει την απόφαση πλαίσιο για τους κρατημένου και αυτή τη στιγμή ε, μόνο ένας με, με δύο έχουν ε, εναλλακτικά μέτρα στην φυλάκιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει ε, διότι κάνουμε αρκετέ συνεδριάσεις με εμπειρογνώμονε, με τα κράτη-μέλη για να τους βοηθήσουμε να μεταφέρουν ε, τα θέματα αυτά. Ε, τον Ιούλιο δημοσιεύθηκε μια έκθεση αξιολόγησης για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη αυτή την απόφαση πλαίσιο και από εκεί και πέρα έγινε και συζήτηση. Να σας δώσω δύο παραδείγματα τα οποία αφορούν το θέμα που αναφέρετε εσείς, το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί υπήκοοι των χωρών. Εάν πρέπει να μεταφερθούν ε, κρατούμενοι ε, με τον τρόπο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, θα υπήρχε δυνατότητα κάποιοι να εκτίσουν την ποινή του στη χώρα καταγωγής τους, στη χώρα που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους και έτσι να ανακουφιστούν κατά κάποιο τρόπο οι υπόλοιποι και να διευκολύνουμε έτσι και την κοινωνική του ένταξη. Ε, τώρα, η απόφαση πλαίσιο για τα μέτρα εποπτείας, το European Supervision Order. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει να το συνθέσουμε με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεστε λόγω του εντάλματος σύλληψης, όχι γιατί πρέπει να εκτίσετε μια ποινή, αλλά γιατί διώκεστε. Εάν εφαρμόσουμε μαζί την απόφαση πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, Σύλληψης και το θέμα της εποπτείας, θα μπορούσαμε ε, πολύ πιο εύκολα να απολευθερώσουμε κάποιον, ιδίω αλλοδαπού, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι, ότι θα τους επιβάλλουμε κάποια μέτρα παρακολούθησης. Για παράδειγμα, ένα ηλεκτρονικό τσίπ ε, στο χώρο διαμονής της. Παραδείγματος χάρη, συλλαμβάνεται ένας Γάλλος, υπάρχει ένταλμα σύλληψη στη Γαλλία, συλλαμβάνεται στο Βέλγιο, μπορεί να επιστρέψει στη Γαλλία ε, ή να μείνει στο Βέλγιο με μέτρα παρακολούθησης ε, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σήμερα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος εν αναμονή της δίκης του είναι υποκράτηση. Δεν απολευθερώνεται. Επομένως αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέτρα ενισχύ τα οποία θα επέτρεπαν να απελευθερώνεται κάποιος ε, πριν, να αποφυλακίζεται κάποιος πριν ε, τη δίκη του και να το επιβληθούν άλλα μέτρα. Και αυτό προσπαθεί να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Να πω και δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, για να απαντήσω λίγο και στη δική σα την ερώτηση, το θέμα των δικαιωμάτων. Όλε οι οδηγίε, οι οποίε ανέφερα στην παρουσίασή μου, παραδείγματο χάρη το θέμα τη διερμηνία και τη μετάφραση, το δικαίωμα στην ενημέρωση, ε, στη πρόταση οδηγία για την πρόσβαση σε συνήγορο ε, συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη και θέλουν να συνεισφέρουν απευθεία στο να ε, βελτιώσουμε τα ελαττώματα του Ευρωπαϊκού Ένταλματο Σύλληψη που παρουσιάσετε στην έκθεσή σα. Παραδείγματο χάρη, στο θέμα τη δίκαιη εκπροσώπηση, του due representation, είπαμε ότι το δικαίωμα πρόσβαση σε συνέργο στην χώρα έκδοση, όχι μόνο στη χώρα εκτέλεση του εντάλματο. Όσον αφορά τώρα και την πρόταση για το γεγονό ότι κάποιο είναι αθώο μέχρι αποδείξει του εναντίον, αυτό και πάλι έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Τώρα, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει. Ε, συνήθως διαβουλευόμαστε την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση ε, επίσημης υπόθεση, Δεν θα το συζητήσω εγώ αυτή σήμερα. Τώρα, η πρόσβαση σε συνήγορο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει ένα φιλόδοξο κείμενο. Είναι οι διαπραγματεύσει εν εξελίξη. Εχθέ έγινε ο τριμερή διάλογο. Συμμετείχα κι εγώ συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι επισήμω πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ενέκρινε τη γενικότερη θέση του Συμβουλίου, έκανε μια συζήτηση με το Κοινοβούλιο και με κάποια κράτη-μέλη για να πει σαφώ ότι για ουσιαστικά θέματα όπω είναι οι παρεκκλήσει και το θέμα του απορρίτου δεν δέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δικαίωμα υπεράσπιση των πολιτών. Εμεί θέλουμε να προχωρήσουμε λοιπόν προ αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε, δεδομένου ότι είναι και διαπραγματεύσει εν εξελίξει, δεν μπορώ να σα πω και περισσότερα. Ε, σα διαβεβαιώ όμω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να έχει ένα φιλόδοξο κείμενο. Αν κατάλαβα καλά τώρα την ερώτησή σα, νομίζω ότι αναφερθήκατε σε δικαστικά ζητήματα τι γίνεται με τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που περιλαμβάνονται στις συνθήκες, ε, ε, δικαιολογούνται σε αυτή την περίπτωση και αν ναι, με ποιο τρόπο. Ωραία. ναι, η νομία δεν είναι αυτή η δικαιοδοσία μου. Γι' αυτό που ρωτήσατε όμως προετοιμάζουμε μια πρωτοβουλία το 2013. Θα δούμε. Είναι Ακόμα είναι νωρίς να πούμε ποια ακριβώς μορφή και περιεχόμενο θα έχει. Νομικό εργαλείο θα είναι πάντως. Ήδη υπάρχει οδηγία όμως σχετικά για την δικαστική αρρωγή. Φαντάζομαι τα απάντησα όλα. Ορίστε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τέλ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπέζε. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο ερώτημα ήδη απαντήσατε. Η Νορβηγία και η Ελβετία δεν αποτελούν τμήμα. Η πρώτη πρόταση της Κομισιόν τους ζήτησε να επιλέξουν εάν το κεκτημένο του Σέγγεν πρέπει να επεκταθεί και στην Ελβετία και Νορβηγία ή αν πρέπει να προβλεφθεί κάτι καινούριο για αυτές τις χώρες και αυτό επιλέξαμε τελικά. Φυσικά υπήρξαν ομοιότητες, αλλά είναι διαφορετική η νομική βάση. Δεύτερον, και πιο αστείο, ε, είναι πολύ φιλόδοξες αυτές οι προτάσεις οι πανμερικοί. Υπήρξαν προσπάθειες να ενδυναμωθούν τα ατομικά δικαιώματα, ε, δικαιώματα της ε, υπεράσπισης, αλλά η συζήτηση βασίστηκε στις εθνικές ποινικέ δικονομίες κάθε χώρας και θα έπρεπε επίσης να προσέξουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση ενός υπόπτου που κατηγορείται σε χώρα άλλη από τη δική του. Και ο κ. Κρόσμπι ανέφερε την εγγύηση να μην δικάζεται κανείς δύο φορές για το ίδιο αδίκημα. Και στο άρθρο 44 του Σέγγεν προβλέπεται αυτό. Είναι πολύ καλό παράδειγμα συγκεκριμένου δικαιώματος σε ένα γενικευμένο χώρο δικαιοσύνης, ασφαλεία κλπ που ξεπερνάει την εθνική ποινική οικονομία και πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση εδώ. Υπάρχουν και άλλα δικαιώματα. Σας ανέφερα ήδη το πρόβλημα της διπλής εκπροσώπησης. Δεν αφορά μόνο εθνική ποινική δικονομία σε μια χώρα μέλος, αλλά και προβλήματα που αφορούν διεθνή επιβολή του νόμου. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι κάποιος που συλλαμβάνεται στη Γερμανία πρέπει να πάει υποχρεωτικά στην Πολωνία και να δικαστεί από πολωνικό δικαστήριο. αυτά δεν είναι αποτελεσματικά. Πρέπει να έχει πρόσβαση και δικαίωμα να εξεταστεί όπως στην Πολωνία. Χρειάζεται λοιπόν ένας νέος μηχανισμός. Και άλλο τώρα. Για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης υπάρχουν και προαιρετικά κριτήρια που δημιουργούν και αυτά κάποια ανισορροπία γιατί οι χώρες μέλη έχουν δικαίωμα να αρνηθούν αν δεν γίνονται σεβαστά θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορούν λέει όμως, μπορούν απλώς. Αυτό πρέπει να αλλάξει και να λέει ότι είναι υποχρεωμένες ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ερήμην. Δεν μπορούμε να εκδώσουμε κάποιον που δεν είναι παρόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα χορηγείται. Είναι εδώ μια έλλειψη προς το παρόν. Μπορούν να αναφερθούν και άλλα παραδείγματα βέβαια, κάποιος να είναι ύποπτος ότι βοήθησε έναν παράνομο μετανάστη ή μετανάστρια. Σύμφωνα με το υπάρχον καθεστώς ισχύει το διπλό κριτήριο. Μέχρι τώρα εξαίρεση χορηγείται σε αυτό μόνο για 32 κατηγορίες αδικημάτων. Νομίζω συμπεριλαμβάνεται και η εμπορία ανηθυρόπων και η αρρωγή σε παράνομους μετανάστες και μετανάστριες, είπατε. Ένα με ότι είναι στον κατάλογο και αυτό. Και στην επεξηγηματική έκθεση εμείς ζητήσαμε αναθεώρησή του. you you can find it there. Okay. Uh, uh, But the second point would be proportionality, hmm. I think. Ναι, υπάρχει και το θέμα της της αναλογικότητας. Δηλαδή, αν είναι να βοηθεί ένα άτομο σε μια περίπτωση, ε, μπορούμε να θέσουμε και το, το ζήτημα της αναλογικότητας εκεί πέρα. εντάξει. θα το επαληθεύσω. Θυμάμαι πω ήταν πρόβλημα όταν ψηφίσαμε την έκθεση. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τι διευκρινήσει σα. Σα ευχαριστώ κύριε Τέλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα στα διάφορα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Οπότε η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 18 Φεβρουαρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και μετά άλλη μια συνεδρίαση στις 19 Φεβρουαρίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30 το απόγευμα. Λίγη τη συνεδρίαση.